Mesdames et messieurs, bonjour. La séance est ouverte. Et je commencerai par euh, quelques annonces. Et la première... Θα ξεκινήσω με κάποιες ανακοινώσεις. Η κυρία Καρολίν Νουκιάς μας ανακοίνωσε το τέλος της θητείας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθότι εξελέγει στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Το σημειώνουμε και σύμφωνα με το άρθρο 7, παραγραφός 2, τις πράξεις όσον αφορά την ε, εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και το άρθρο 4, παράγραφος 4 ανακοινώνουμε ότι η θέση της είναι κενή από την 18 Μαΐου 2010. Από τις 12 Μαΐου ο κύριος Μακμίλαν Σκοτ ανήκει στην ομάδα των φιλελευθέρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορούμε να περάσουμε αμέσως τώρα στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Θα ξεκινήσω αμέσως με την έκθεση Μαλκά. Πρόκειται για τον διορθωτικό προϋπολογισμό 01-2010 και κατόπιν έκθεση Τρίπελ όσον αφορά τις προβλέψεις για τα έσοδα και τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2011. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Βλάντιμιρ Μάνκα για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ. Βάσει τη συνθήκη τη Λισαβόνα, ξέρετε ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα που γίνονται σαφέστερα και πιο διαφανή. Υπάρχει ένα καλύτερο ορισμό των αρμοδιοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε περισσότερε αρμοδιότητε και βεβαίως ε, αποκτήσαμε νέες αρμοδιότητες. Για πρώτη φορά οι πολίτες περισσότερων χωρών έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν με κάποιο τρόπο τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη και θα ήθελα επίσης να πω ότι όλοι οι πολίτες ακόμα και αυτοί που βρίσκονται πιο μακριά από τα κέντρα εξουσίας έχουν δημοκρατικά μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Αυτά τα δημοκρατικά μέσα και εργαλεία βεβαίως δεν θα πρέπει να επιβαρυνθούν με σημαντικά οικονομικά μέσα. Η Συμφωνία της Λισαβόνας, η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει συγκεκριμένες ε, επιπτώσεις και για το 2010 υπάρχει μια συμφωνία η οποία ορίζει το περιθώριο ελιγμού για το τμήμα 5 καθώς και για τη χρηματοδότηση αυτών των επιπλέον δαπανών. Από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία της Λισαβόνας χρειάστηκε να συζητηθεί αυτή η επιπλέον επιβάρυνση αυτός ο διορθωτικός προϋπολογισμός. Έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης των προβλέψεων, έχοντας υπόψη το περιθώριο ελιγμού το οποίο έχουμε και βεβαίως κοιτώντας προηγουμένως πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες αυτές δαπάνες μέσω των υφιστάμενων δημοσιονομικών μηχανισμών και πόρων. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε και την δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίξει το ρόλο του σαν συνομοθέτη. Οι συγκεκριμένες επιπτώσεις λοιπόν στον πραγματικό προϋπολογισμό είναι χαμηλότερες από αυτές που αρχικά είχαν προβλεφθεί. 4 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό οι επιπλέον αυτές δαπάνες. Καταρχήν λοιπόν θα προσπαθήσουν να προκύψουν και από εξοικονομήσεις και αναδιάταξη των υπάρχοντων πόρων. Υπάρχει επίσης και αυτός ο μήνας διαφορά μεταξύ της αρχικής συζήτησης και της απόφασης. Η οικονομική κρίση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ε, οικονομίας. Πιστεύω ότι αυτό ισχύει όχι μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω εξοικονομήσεις, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, όχι μόνο για το 2010 αλλά και για τα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο εξαρτάται από το Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μεγάλο βαθμό. Οι αποφάσεις αυτές οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι οι συζητήσεις και η συνάντηση που θα καταλήξει το Δεκέμβριο μπορεί να μας οδηγήσει σε περαιτέρω εξοικονομίες. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Η κυρία Τρούπελ έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Η συγγήτρια. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, για το 2011 για πρώτη φορά έχουμε ένα σωστό προϋπολογισμό σωστό μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκη τη Λισαβόνα, Έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες, έχουμε περισσότερα καθήκοντα, έχουμε περισσότερες ευθύνες, έχουμε περισσότερες ευθύνες και αρμοδιότητες στον νομοθετικό τομέα περισσότερη δυνατότητα εργασίας, άρα χρειαζόμαστε και περισσότερα δημοσιονομικά μέτρα. Την ίδια ώρα θα πρέπει να δούμε η οικονομική κρίση, η σταθερότητα του ευρώ η κρίση που θα οδηγήσει σε όλες τις χώρες αλλά και στη Γερμανία σε σημαντικές ε, αναδιαρθρώσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε και την Ελλάδα και τα άλλα υπερχρεωμένα κράτη. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε υπεύθυνοι στη στάση μας σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση και να προχωρήσουμε σε κάποιες σημαντικές αλλαγές στον προϋπολογισμό του 2011. Σαν εισηγήτια Προσπάθησα να στηρίξω την θέση των περισσότερων, αλλά θα προσπαθήσω να σας μιλήσω και για τη θέση των πρασίνων. Όσον αφορά το διοικητικό προϋπολογισμό, έχουμε το ανώτατο όριο, το οποίο έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών του Κοινοβουλίου και των διαφόρων συζητήσεων έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες, έχουμε περισσότερες ευθύνες και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πάρουμε ακραίες θέσεις. Χρειάζεται αυτοπιθαρχία, χρειάζεται περισσότερη <clears throat> αυτοπιθαρχία για να παραμείνουμε σε αυτό το 20%. 4,6% επιπλέον δηλαδή πάνω από τα 13 εκατομμύρια τα οποία ήδη έχουν ε, αποφασιστεί για το 2010, συμφωνήσαμε ότι αυτό το 20,28% δηλαδή πάνω από 20 εκατομμύρια είναι το ποσό το οποίο δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε. Επίσης περισσότερες θέσεις για την πληροφορική, για τη βιβλιοθήκη, για τις έρευνες, για την εμπειρογνωμοσύνη τομείς για τους οποίους χρειάζεται η στήριξη όλων των ειδικών έτσι ώστε να μην ε, επιβαρύνουμε περαιτέρω το υπάρχον προσωπικό. Πού υπάρχουν όμως ε, έντονες συζητήσεις για το 2011. Υπάρχουν παραδείγματο χάρη τα ποσά για τους βοηθούς. Όχι για τα μέλη του Κοινοβουλίου, αλλά για τους βοηθούς 13,2 εκατομμύρια ευρώ. Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, αυτή η συζήτηση πρέπει να σας πω δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, τα περισσότερα λοιπόν μέλη της Επιτροπής θεώρησαν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για το ποσό αυτό. Οι πράσινοι, πρέπει να σας πω, ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, θεωρούν ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί η πολιτική μου ομάδα λοιπόν θεωρεί ότι αυτή η αύξηση των 1.500 ευρώ, ποσά επαναλαμβάνω που είναι μόνο για τους βοηθούς, θα πρέπει να μην εγκριθούν. Θεωρούμε ότι θα πρέπει για το επόμενο τουλάχιστον έτος να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, κάτι το οποίο και από πολιτικής απόψεως έχει περισσότερη βαρύτητα. Να είμαστε λοιπόν πιο αποτελεσματικοί. Αυτό το 12,9% περιορισμό των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα είναι ένας από τους στόχους καθώς και η βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα. Θέλουμε να μειωθούν οι περιβαλλοντολογικές μας επιδόσεις και αυτό είναι ένας από τους στόχους στους οποίους δεν θα υποχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τρίπελ, εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Φερνάντες έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υποστηρίζει σαφώς την διαφάνεια και την βιωσιμότητα του προϋπολογισμού. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πολύ θετικό το έργο που έχει ε, πληρώσει η διοίκηση για να αποφασίσει τις πάγιες και μεταβλητές δαπάνες μας, παρουσιάζοντας και μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την πολιτική ακινήτων. Ωστόσο, θεωρούμε ότι το κείμενο αυτό θα μπορού, τα κείμενα αυτά θα μπορούσαν να βελτιωθούν στο μέλλον. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε προτείνει μια στρατηγική μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για τα ακίνητα. Σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των δαπανών, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς έναν μηδενικό προπολογισμό, έναν προπολογισμό που θα ξεκινά από μηδενική βάση για να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε την, μια, μια ευρύτερη σωστή προσέγγιση βάσει μιας ανάλυσης κόστους όφελους κάθε ε, δαπάνης. Ε, υποστηρίζουμε τις ε, περικοπές των δαπανών και τις μειώσεις σε κάποιες κατηγορίες. Ε, η νομοθετική επιτυχία πρέπει να είναι ο στόχος του Κοινοβουλίου. Όλοι γνωρίζουμε ότι το... η, η μη ύπαρξη νόμου ή ένας κακός νόμος έχει υψηλό κόστος που εν τέλει έχει επίπτωση στους Ευρωπαίους πολίτες. Για να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις που προκύπτουν από τις νέες αρμοδιότητες που έχουμε μετά την έναρξη τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη της Λισαβόνας και για να πετύχουμε την νομοθετική αριστεία που θέλουμε, θέλουμε να υπάρξουν νέοι ανθρώπινοι πόροι που πρέπει να είναι υψηλή ποιότητα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι θα έχουμε 18 νέους βουλευτές που πρέπει να έχουν τις απαραίτητες ε, προϋποθέσεις για να ασκήσουν επιτυχώς τις αρμοδιότητές τους. Ζούμε μια απαιτητική στιγμή, κατά την οποία τα ευρωπαϊκά όργανα καλούνται να παίξουν έναν καθοριστικό σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας επαρκή μέσα. Γνωρίζουμε ότι σε θέματα προϋπολογισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί έντονα λαϊκισμός δημαγωγία. Αυτό το απορρίπτουμε. Κάποιοι αφήνουν να, υπο, να υπονοηθεί ότι αυξάνονται οι δαπάνε για του βουλευτέ. Αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Αυτό που ζητούμε είναι να υπάρχουν επαρκεί πιστώσει, ούτω ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λειτουργεί με αξιοπρέπεια όπω όλοι ζητούμε και να πετύχει το στόχο που προσδοκά ο Ευρωπαίο πολίτη που απαιτεί ο Ευρωπαίος πολίτης από εμά την ε, νομοθετική αριστεία. Ευχαριστώ κύριε Φερνάντε. Ο κύριος Βόγκαν έχει το λόγο για τρία λεπτά. Πάντοτε ε, υπάρχει μια σύγχυση κάθε φορά που συζητούμε τον προϋπολογισμό και ε, το ίδιο ισχύει και με τον διορθωτικό προϋπολογισμό. Πάντως χαίρομαι που τα περισσότερα θέματα έχουν επιληθεί από την ίδια την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Και τώρα υπάρχουν ελάχιστες διαφορές μεταξύ των θέσεων της Επιτροπής Προϋπολογισμών και του Προεδρείου εκτός από τρία θέμα, τρία, τέσσερα θέματα. Το ένα είναι το όριο του 20%, το δεύτερο τα αποθεματικά και ε, το, το άλλο είναι τα 1.500 ευρώ μηνιαίως για τους βοηθούς. Αυτά τα 1.500 ευρώ πράγματι είναι ένα επίμαχο θέμα το οποίο θα συζητηθεί και ιδιαίτερω σε εποχές οικονομικά δύσκολες. Και παρά το γεγονός ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας μας έχει δώσει νέες ε, ευθύνες και αρμοδιότητες. Τώρα, σχετικά με την χρηματοδότηση του δεύτερου γύρου αυτών της διάθεσης των 1.500 ευρώ ε, σε ένα αποθεματικό είναι πιο λογική ε, προσέγγιση. Ένα άλλο επίμαχο θέμα είναι το ειδικό ποσό για την διατήρηση του, των γραφείων. Εδώ έχουμε ένα συνολικό ποσό 400.000 ε, ευρώ και κάθε φορά που ε, δαπανάτε ε, ποσό σχετικό με αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να υπάρχει ειδική τεκμηρίωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, δεν ξέρω αν οι δύο αυτές συμβαστικές λύσεις είναι αποδεκτές ή όχι. Ελπίζω ότι η πλειοψηφία θα τις δεχθεί. Ωστόσο, ένα άλλο πράγμα κατέστη σαφές στις ε, συζητήσεις μας για τον προϋπολογισμό του 2011. Δηλαδή, αν είναι να χρηματοδοτήσουμε επιπρόσθετες ε, αρμοδιότητες, σύμφωνα με την συνθήκη της Λισαβόνας, θα πρέπει ταυτόχρονα να αναζητήσουμε και εξοικονομήσεις από κάποιους άλλους ε, τομείς. Πράγματι έχουν γίνει σημαντικές εξοικονομήσεις και ε, η συνολική αύξηση μειώνεται από 6,5% σε 5,8%. Χαίρομαι γι' αυτό και ελπίζω ότι το Προεδρείο θα προτείνει συστάσεις και ε, προτάσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να κάνουμε αποτελεσματικές εξοικονομήσεις στο μέλλον. Παραδείγματος χάρη αλλαγή στον τρόπο που κάνουμε πράγματα και όχι απλώς να κάνουμε περικοπές. Ελπίζω ότι αυτή θα είναι η στάση μας στο μέλλον αφού το θέμα συζητηθεί με τα μέλη ε, εγκαίρως. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, μοιραστεί τις θέσεις και απόψεις του ε, με όλους και να δώσει απαραίτητες εξηγήσει. Ταυτόχρονα ο προϋπολογισμός μας θα πρέπει να είναι απολύτως αποδεκτός τόσο στα μέλη του Κοινοβουλίου όσο και στο κοινό. Ευχαριστώ. Ο κύριο Άγνουντς έχει το λόγο τώρα για τρία λεπτά εκ μέρους των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η κυρία του έκανε πολύ καλή δουλειά όταν προσπάθησε να παρουσιάσει έναν πιο ισορροπημένο από τον αρχικό προπολογισμό. Είναι σαφές ότι η συνθήκη της Λισαβόνας θέτει νέες προκλήσεις και νέες αρμοδιότητες για όλους μας και άρα θα έχει υψηλότερο κόστος. Η πρόταση προσπαθεί να ισορροπήσει τις αντιμαχόμενες αυτές θέσεις. Εμείς δεν μπορούμε να αναδιοργανώσουμε τη δουλειά, τον τρόπο δουλειά μας σε επίπεδο συνεδριάσεων, οπότε και σε πολλά διοικητικά θέματα. Κάλιστα ωστόσο θα μπορούσαμε εκεί να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ε, όπως αναφέρθηκε, ε, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι νέες δυνατότητες που μας προσφέρουν οι τεχνολογίες και οι ανάγκες περικοπών. Η αύξηση των 1.500 ευρώ για κάθε ευρωβουλευτή σε ό,τι αφορά τις, ε, την αμοιβή των συνεργατών τους είναι κάτι θετικό. Πιστεύω ωστόσο ότι αυτό θα έπρεπε να λειτουργήσει και σε επίπεδο επιτροπών είναι σαφές ότι πρέπει να δουλέψουμε στις ομάδες για να δούμε πώς μπορούμε να ε, το επεξεργαστούμε καλύτερα. Είναι σαφές ότι αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει μια καλύτερη, ένας καλύτερος τρόπος δουλειάς περιορίζοντας τις δαπάνες σε μια λογική ωστόσο που ε, δεν θα οδηγεί σε μείωση της απόδοσής μας. Αυτό ε, πρέπει να το δούμε και σε νούμερα και σε απόδοση. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν συνεργάτες που δουλεύουν και αυτοί εδώ και πρέπει να προσπίζουμε τις συνθήκες δουλειά τους. Νομίζω ότι εν γέννη μπορούμε να το δούμε επικριτικά με χωρίς ωστόσο να αγνοούμε τα θετικά του στοιχεία. Κυρία Τρίπελ, 1,5 λεπτό για τους πράσινους. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτή τη μαγική λέξη, ισορροπία που ανέφερε ο τελευταίος ομιλητής. Όταν μιλάμε για το 2011, στις ε, συζητήσεις και διαβουλεύσεις που είχαμε, προσπαθήσαμε να δούμε πού είναι αυτό το σημείο ισορροπίες για να προσανατολιστούμε προς τα εκεί. Μίλησε για λαϊκισμό ο συνάδελφος. Εγώ πιστεύω ότι προσπαθήσαμε πραγματικά να δείξουμε υπευθυνότητα και αυτοπιθαρχία όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2011. Θα πρέπει όλοι, πιστεύω, να συνειδητοποιήσουμε πόσες εξοικονομήσεις είναι απαραίτητες. Αυτά που απαιτούμε από κάποια κράτη να τα επιβάλλουμε και στον εαυτό μας. Αυτό δεν είναι λαϊκισμός. Αυτό κατά την άποψή μου είναι πολιτική υπευθυνότητα που δείχνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη σημερινή κατάσταση όταν ζητάμε και απαιτούμε από την Ελλάδα τέτοιους τρομερούς περιορισμούς και περικοπές θα πρέπει να έχουμε και εμείς το θάρρος να επιβάλλουμε τις αντίστοιχες περικοπές και εξοικονομήσεις στον εαυτό μας και να βρούμε την ίδια ώρα και ένα όριο όπου να πούμε ότι στην σημερινή κατάσταση θα πρέπει να υπάρξει ένα ανώτατο όριο. Ανήκουμε και εμείς στο ίδιο πολιτικό περιβάλλον και έχουμε συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει γύρω μας. Γι' αυτό και κάνω μια έκκληση προς όλες τις πολιτικές ομάδες να συνειδητοποιήσουν τι μήνυμα στέλνουμε στην κοινή γνώμη με αυτό τον προπολογισμό 2011. Ευχαριστώ κύριε Τρούπελ. Ο κύριος Πόκοδος, δύο λεπτά, για τους μεταρρυθμιστές και συντηρητικούς. στην Ρουμανία υπάρχει περικοπή 25% των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Στην Ισπανία 5 με 25% των μισθών των υπαλλήλων χάνονται. Στην Πορτογαλία, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, οι κυβερνήσεις κάνουν τεράστιες προσπάθειες για να μειώσουν τους πόρους. Η νέα κυβέρνηση στη Μεγάλη Βρετανία ανέφερε ήδη την ανάγκη μείωση ε, μεγάλων περικοπών. Στο κοινοβούλιο όμως πιστεύει κανείς ότι είναι καιρό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αρχίσει να ξοδεύει οτιδήποτε περισσότερο οπουδήποτε σε οποιαδήποτε ε, ε, σε οποιοδήποτε θέση του προπολογισμού, προσωπικό, ε, γραφεία, βιβλιοθήκες, 1.500 ευρώ για αύξηση των επιδοτμάτων των συνεργατών των βουλευτών. Είναι παράλογο και περιττό. Το δεύτερο λοιπόν, ήδη ο πρώτος ε, διορθωτικός υπολογισμού είναι υπερβολικός, πόσο μάλλον ο δεύτερος. Δεν είναι καιρός να ε, κάνουμε κάτι τέτοιο. Ξέρουμε ότι, χρειάζονται, ότι περισσότεροι, έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες, αλλά αυτό δεν απαιτεί περισσότερες δαπάνες, αλλά αποτελεσματικότερες δαπάνες, μεγαλύτερη λογοδοσία και μεγαλύτερη ευθύνη. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Τρίπελ όταν είπε ότι υπάρχουν δυνατότητες επιπρόσθετων ε, περιορισμών. Δεν χρειαζόμαστε και άλλα αυτοκίνητα. Υπάρχει δωρεάν, ε, δωρεάν δυνατότητα μεταφοράς μας με, με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Εγώ έχω μια κάρτα, ε, έχω μια κάρτα με τα μέσα ενημέρωση, με τα μέσα μεταφοράς με τα οποία επιτρέπουν να ταξιδεύω συνεχώς. Όλοι γνωρίζουμε λοιπόν ότι οι συζητήσεις μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προπολογισμών ήταν χρήσιμες. Ωστόσο, εγώ βλέπω ότι έχουμε πολύ περισσότερες ακόμα ευκαιρίες μείωση των δαπανών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Άντρεσεν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για μία ακόμα φορά με μένω εμβρόντετη πως οι αριθμοί στο πλαίσιο αυτού του προϋπολογισμού διονγκώνονται ενώ οι λαοί υποφέρουν από την οικονομική κρίση. Σήμερα όμως θα αναφερθώ στην ηθική αυτού του Κοινοβουλίου. Υπό την παρούσα κατάσταση είναι αποδεκτό ενώ ζητούμε περιορισμό των εθνικών δαπανών τα ευρωπαϊκά όργανα να αυξάνουν τον προϋπολογισμό στα διοικητικά. Είναι αποδεκτό τα θεσμικά όργανα να προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όταν ε, ζητάτε να υπάρξει κάποια ε, κάποιος περιορισμός στους μισθούς ε, των, ε, των υπαλλήλων των ευρωπαϊκών οργάνων. Είναι λογικό το Κοινοβούλιο να δέχεται τους λογαριασμούς του 2008 του Συμβουλίου όπου είχε επιφυλάξει σε αντάλλαγμα της έγκρισης του παρόντος προϋπολογισμού. Δυστυχώς, τότε είχαμε καταγγείλει το Συμβούλιο για έλλειψη διαφάνειας. Συμπτωματικά το Συμβούλιο ε, δεν συμφώνησε με τις αυξήσεις του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου. Ε, όλα αυτά πρέπει να δημοσιοποιηθούν αμέσως μετά ε, το Συμβούλιο θα εγκρίνει το πρόσθετο προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η εικόνα της Ευρώπης. Δηλαδή, ε, ο εκπρόσωπός μας επιθεμάτων θεμάτων δεοντολογίας ε, θα πρέπει να δει πώς θα ε, διέπει η δεοντολογία όλους μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Βέρτμαν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμοι συνάδελφοι. Συμφωνία της Λισαβόνας ε, οδήγησε σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την οργάνωσή του. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι απαραίτητο να διορθωθεί. Βεβαίως και τίνουμε όλοι προς την αριστεία, προς την βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία. Το θέμα όμως είναι ότι βρισκόμαστε εν μέσω της σοβαρότερης οικονομικής κρίσης τα τελευταία 60 χρόνια. Και αναρωτιέμαι εμείς σαν Ευρωπαίοι βουλευτές μήπως θα πρέπει να δείξουμε τρομερή προσοχή, πολύ μεγαλύτερη προσοχή τουλάχιστον από αυτή που δείχνουμε μέχρι τώρα όσον αφορά την δαπάνη, όσον αφορά τη λειτουργία και όσον αφορά την οργάνωση του ε, οργάνου μας εδώ.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 θα πρέπει να είμαστε υπόδειγμα ε, τιμιότητας καθώς δαπανούμε τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών. Από την άλλη όμως θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να εκπληρώσει όλες του τις ε, υποχρεώσεις σύμφωνα με τη συνθήκη της ε, ε, Λισαβόνας. Είναι αληθές ότι σύμφωνα με τη νέα συνθήκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει ένα ε, σημαντικό μερίδιο ευθυνών. Δική μας υποχρέωση είναι να τηρήσουμε τις παραδόσεις της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και να συμβάλλουμε ώστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητα του Κοινοβουλίου και να διατηρήσουμε την καλή του ε, φήμη. Οι συζητήσεις οι οποίες έγιναν δείχνουν σε ποιο βαθμό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη ε, τι ε, δυσχερείς οικονομικές συνθήκες και λαμβάνει ανάλογες αποφάσεις. Η συζήτηση ακριβώς αντανακλά την οικονομική κατάσταση. Αυξήσαμε το κόστος κατά 5,5%. Δίνουμε το παράδειγμα ε, περιορίζοντας ε, περιορίζοντας ε, όλες τις δαπάνες και αυξάνοντας μόνο κατά 20,8% τις νέες δαπάνες σύμφωνα με την συνθήκη. Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν όλες αυτές οι βασικές αρχές δεδομένων των νέων αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο μέλλον θα πρέπει να καταβάλουμε πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του έργου του Κοινοβουλίου ε, δίδοντας την έμφαση όχι στα κτίρια αλλά στις νέες τεχνολογίες και να δώσουμε και το παράδειγμα τόσο ως προς την προστασία του περιβάλλοντος ε, και τη λειτουργία των ε, κτίριων. Σε καμία περίπτωση ο προπολογισμό δεν θα πρέπει να διονγκώνεται αυτομάτω, κάτι το οποίο αρέσει στι στις Ο κύριος Αλβάρο έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Herzlichen Dank. Ich glaube, besonders in Krisenzeiten müssen Politiker in der Lage sein, Rationalität und Emotionalität voneinander zu trennen, besonders wenn wir über Haushaltsfragen und Geld sprechen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 και καλείται να διαδραματίσει ένα σημαντικότερο ρόλο μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, θα πρέπει για το σκοπό αυτό να έχει τα απαραίτητα ε, χρηματοδοτικά μέσα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πράξη. Είναι βέβαιο όμως ότι θα διευρυνθεί το πεδίο της δράσης μας και άρα και οι προσδοκίες από πλευράς των πολιτών θα αυξηθούν. Συνεπώς, η πρόταση για αύξηση ε, της αμοιβή των ε, βοηθών πολιτικά αλλά και γενικότερα είναι δικαιολογημένη. Ε, βεβαίως όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μια σοβαρή κρίση στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Ωστόσο, δεν, δεν μπορούμε να ε, ε, να δημιουργήσουμε δυσλειτουργία σε κάποιες από τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάνοντας περικοπές. Γι' αυτό λοιπόν είναι απολύτως δικαιολογημένη αυτή η αύξηση. Ο κύριος Βάντερ Στούπ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2011 συνολικά καλύπτει 1,7 δις ευρώ. 600 ευρώ την ημέρα για κάθε βουλευτή. Μιλάμε για αρκετά χρήματα. Και αναρωτιέμαι τι μπορούμε να κάνουμε για να, για να χρηματοδοτήσουμε κάτι άλλο και όχι το, αυτό το παιχνίδι. Θα έπρεπε να σταματήσει αυτό το πήγαινέλα μεταξύ Βρυξελών, Στρασβούργου, Λουξεμβούργου. Ένα τμήμα του προπολογισμού πρέπει να το ξαναγυρίσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες που υποφέρουν στην καθημερινότητά τους από τις περικοπές. Πώς να εξηγήσουμε στον Ευρωπαίο φορολογούμενο ότι η γραμματεία θα, κάθε γραμματέας ευρωβουλευτών θα στοιχίζει 1500 ευρώ το μήνα περισσότερο ενώ, αυτός, ενώ από αυτόν θα πρέπει να κόψουμε μισθούς. Ε, θέλουμε στο Κοινοβούλιο και άλλα και άλλα και άλλα. Υπάρχουν όμως συμφωνίες που γίνονται στους διαδρόμους και, και κλεισμένων των θυρών που δεν ξέρει κανένας αλλά που πληρώνει ο φορολογούμενος. Θα ήθελα σήμερα να ξανασκεφτούμε το κόστος των αυξήσεων για κάθε βουλευτή, για κάθε μέρα. Αυτό και μόνο θα ήταν ένα θετικό. Η κυρία Γκρέσλε, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί. Κύριε Βαντιστόπ, εγώ μετράω με μεγάλη προσοχή τις δαπάνες και θεωρώ ότι έχουν αξία τα χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου. Πιστεύω λοιπόν ότι ακριβώς επειδή οι δαπάνες που προτείνονται θα δημιουργήσουν και κάποιες επιπλέον θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει να κοιτάξουμε με προσοχή τι προτείνουμε. Εδώ προτείνουμε επιπλέον θέσεις απασχόλησης για να εργαστεί αυτό το κοινοβούλιο με ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τρόπο. Χρειαζόμαστε κάποιους συνεργάτες. Αν δεν τους χρειαζόμαστε και μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς, τόσο το καλύτερο. Αλλά εγώ πολύ φοβάμαι ότι αν θέλουμε άτομα αξιόλογα, τα οποία να υποστηρίζουν την εργασία μας, θα πρέπει να τους πληρώνουμε ικανοποιητικά και θα πρέπει να έχουμε ικανό αριθμό. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε κατά πόσο είναι δικαιολογημένε αυτές οι δαπάνες, αυτές οι επιπλέον θέσει και αυτές οι δραστηριότητε. Υπάρχουν πράγματα που σαφώς μπορούν να ξεχαστούν όπως ε, τα ποσά που προτείνονται για κάποιες νέες τεχνολογίες, ε, για την κινητή την εφολία. Όμως υπάρχουν τομείς για τους οποίους πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βανόρντεν για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, σε ολόκληρη την Ευρώπη οι κυβερνήσεις και τα δημόσια όργανα ε, προχωρούν σε περικοπές. Δυστυχώς αυτό το κοινοβούλιο ζει σε ένα παραμυθένιο κόσμο. Ε, ακούμε τα λόγια, ακούμε όρους όπως εξοικονόμησης και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, ο διορθωτικός προπολογισμό ε, προβλέπει μια αύξηση 6% για τον προπολογισμό του 2011. Δεν γίνονται εξοικονομήσει λοιπόν. Θα μπορούσαν να γίνουν αρχίζοντα από το προσωπικό με άχρηστε δαπάνε. Ε, θα πρέπει να δώσουμε ένα τέλος στο τσίρκο τόσο του Συμβουλίου όσο και του Στρασβούργου με μια πολύ σημαντική ε, μείωση 50 εκατομμύρια ευρώ κλείνοντας τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάθε μία από τις χώρες μας να υπάρξει περικοπή της γραφειοκρατίας ο αριθμός των ε, υπαλλήλων αυξάνει κατά 14% από το 2004 και εντεύθυνα χρειάζεται να τεθούν ε, νέες προτεραιότητες ε, με περικοπές δαπανών. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο κυρία Πρόεδρε και πρέπει να ε, κάνουμε πολύ σοβαρά και σημαντικά βήματα για νέες περικοπές και μειώσεις στο προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ και τώρα περνούμε στις ελεύθερες παρεμβάσεις και το λόγο έχει ο κύριος Στάς. Eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Θα ήθελα να μιλήσω για τα επιπρόσθετα 1.500 ευρώ για τα έξοδα γραμματείας. Είναι γεγονός ότι η Λισαβόνα επιβάλλει νέες δουλειές, νέα καθήκοντα. Εγώ δεν είμαι αντίθετο στο να υπάρχουν περισσότεροι περισσότερα μέλη προσωπικού στις γραμματείες των επιτροπών που έχουν περισσότερες αρμοδιότητες, όπως την Επιτροπή Γεωργίας. Ούτε διαφωνώ με την ένταξη περισσότερων υπαλλήλων στις ομάδες, για να δουλεύουν σωστότερα οι ομάδες. Θα ήθελα ωστόσο να πω ότι το να παίρνουν κάθε βουλευτής επιπλέον 1500 ευρώ το μήνα είναι παράλογο αυτή τη στιγμή. Εγώ δούλεψα 10 χρόνια στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που έχει πολλά νομοθετικά καθήκοντα, πολλές ευθύνες, πολλά θέματα που ανήκουν στην απόφαση και έχω να, συνεχίζω να έχω τρεις συνεργάτες. Οι συνάδελφοι που δουλεύουν στην γεωργία ή τις δημόσιες ελευθερίες μπορούν και αυτοί να καλύψουν τη δουλειά τους με τρεις. Κύριε Γκρέσλε, αυτοί που θέλουν να δουλεύουν ε, δεν σημαίνει ότι αυτοί που θέλουν περισσότερο προσωπικό θέλουν να δουλεύουν περισσότερο και οι άλλοι όχι. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι ο λαϊκισμός δεν υπάρχει κανείς άλλος στη διαδικασία του Catch the Eye. Δίνω ξανά το λόγο λοιπόν στους δύο σου εισηγητές, τον κύριο Μάνκα. Καταρχάς, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους παρουσίασαν τις απόψεις τους και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί οι απόψεις ε, όλων συγκλίνουν ότι πρέπει να οργανώσουμε καλύτερα τις εργασίες μας και να τίνουμε προς περισσότερη εξοικονόμηση και αποτελεσματικότητα. Ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά νομίζω ότι όλοι συμφώνησαν σε αυτό. Ο κ. Μπόκρος είπε ότι υπάρχουν αντικειμενικές εξοικονομήσεις και περικοπές. Αυτός είναι ο τρόπος που πριν από ένα χρόνο απέρριψαν ε, τα μέλη της πολιτικής του ομάδας. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά την κοινή γνώμη και όσον αφορά την ε, εντύπωση που δίνουμε προς τα έξω, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να μας καθοδηγήσει όσον αφορά τις ε, εξοικονομήσεις που θέλουμε να κάνουμε. Η καλύτερη οργάνωση, η αναδιάρθρωση των ε, υπαρχουσών δυνατοτήτων, η καλύτερη χρησιμοποίηση των υπάρχοντων μέσων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο καλύτερος τρόπος για να περικόψουμε τα έξοδα και τις δαπάνες μας. Περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία την Επιτροπή Περιφερειών αλλά και την ε, Οικονομική ε, Επιτροπή, καθότι οι δικές τους ψηφοφορίες σαφώς και θα δώσουν και ένα μήνυμα. Η έκκληση μου είναι να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό έτσι ώστε να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει τις νέες του αποστολές και τις νέες του αρμοδιότητες. Η κυρία Τρίπελ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ακούσατε όλοι ότι υπάρχει αντιπαράθεση για τον προεπολεσμό 2011. Πολλές και διαφορετικές απόψεις. Από τη μία υπάρχει η εξοικονόμηση, οι περικοπές. Από την άλλη έχουμε μια συμβολική πολιτική και ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να στείλουμε προς τα έξω. Είδατε, ακούγοντας την κυρία Κρέτσι το ΕΛΚ, τι ε, απόψεις έχει όσον αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών και τους συνεργάτες που χρειαζόμαστε για να διεκπαιρεώσουμε τις αποστολές μας. Και ακούσατε και άλλους συναδέλφους οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει όλα αυτά να καταργηθούν και να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε με λιγότερα μέσα και λιγότερο προσωπικό. Η πλειοψηφία όμως της Επιτροπής συμφώνησε αυτά τα επιπλέον πώς να μπουν στο αποθεματικό δεν έχουν αποφασίσει δηλαδή να τα καταργήσουν, ζήτησαν όμως μια καλύτερη αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών. Αξιολόγηση η οποία θα πρέπει να υποβληθεί με αριθμούς, με στοιχεία δικαιολογημένη και το φθινόπωρο να συνεχίσουμε τη συζήτηση τον Οκτώβριο με τη νέα διαδικασία του προπολογισμού και με το Συμβούλιο να συνεχίσουμε τη συζήτηση καθώς και εδώ στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε μια δυνατή πλειοψηφία. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των μεν και των δε, αλλά υπάρχει και μία θέση της πλειοψηφίας η οποία θέση της πλειοψηφίας είναι περαιτέρω εκτίμηση και αξιολόγηση αυτών των αριθμών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Τρίπελ. Έτσι ολοκληρώνεται η κοινή συζήτηση για το προϋπολογισμό. Ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις τους. περίπου η συζήτηση. Η